So, dear ladies and gentlemen, would like to continue. Κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δικαιωμάτων Γενικών και Ανάπτυξης. Είναι το σημείο 9 της σας διαταξης διάταξης. 20η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη ή συντομότερα Σύνοδος Κορυφής του Ναϊρόμπι. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα βεβαίως να καλωσορίσω τον ε, συμπρόεδρό μου, τον κύριο Τομπέ, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Θα μιλήσουμε αρκετά θα μιλήσω εγώ και στη συνέχεια θα, θα συνεχίσει ο κύριος Τομπέ. Γιατί, γιατί ε, θέλουμε βεβαίως να εμφανιστούμε εδώ με τις διάφορες ιδιότητές μας και ως πρόεδροι των Επιτροπών αλλά και ως ε, συντάκτες των, ε, του σχεδίου ε, ψηφίσματος που θα κατεβάσουμε στην, στην, στην Σύνοδο Κορυφής του Ναϊρόμπι που θα ε, συνοδεύει και μια προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν εν ώψη της ε, Συνόδου Κορυφής. Έχουμε ήδη συντάξει ένα τέτοιο κείμενο που θα είναι η αφετηρία μας για τις συζητήσεις ε, που θα έχουμε με διάφορους παράγοντες ε, ε, το επόμενο διάστημα εν ώψη της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής. Βεβαίως θα πρέπει από γενική άποψη να προσέξουμε και να προετοιμάσουμε πολύ καλά την Σύνοδο Κορυφή αυτή. Πρέπει να δώσουμε προσοχή σε διάφορα σημεία. Γι' αυτό και είπα ότι θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω από ό,τι ήθιστε. Θα δώσω το λόγο και στο συμπροεδρό μου και θα σας παρουσιάσουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Το σχέδιο κειμένου θα σας το παρουσιάσουμε και οι δύο, εγώ και ο κύριος Τομπέ με, ε, ως, πρόεδρο, ως πρόεδροι και εισηγητέ των δύο επιτροπών μας. Ξέρετε ότι η Σύνοδος του Ναϊρόμπι ε, γίνεται 25 χρόνια μετά την ε, αντίστοιχη Σύνοδο Κορυφής του Καΐρου που αποτέλεσε ένα τεράστιο ορόσημο οπότε 179 χώρες ε, ανέλαβαν δεσμεύσει για την καταπολέμηση ε, προβλημάτων που υπήρχαν όσον αφορά την σεξουαλική ε, και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και την κατάρτιση ενό θεματολογίου για την ισότητα των φίλων. Η σύνδεση Κορυφή αυτή αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να επανεπιβεβαιώσουμε τις δεσμεύσει κυβερνήσεων και κρατών στην ε, ε, εξάλληψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την ε, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Στο ψήφισμα λοιπόν καταγράφεται και η προοδός που έχει σημειωθεί, η αύξηση της διαθεσιμότητας μέσων αντισύλληψης και η μείωση της βρευκής θνησιμότητας. Όμως τονίζει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες αν θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος όσον αφορά ε, την αυτοπραγμάτωση του μισού πληθυσμού του πλανήτη. Όσον αφορά το, την πρώτη δέσμευση της ε, Συνόδου Κορυφής του Ναϊρόμπι, όσον αφορά τον οικογενειακό σχεδιασμό, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ζητούμενο μόνο η διαθεσιμότητα, αλλά και η πρόσβαση στις υπηρεσίες. Και θα πρέπει να ε, εξασφαλίζεται επίσης, πέρα από τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει να καλύπτει όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, ε, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ε, από το αν πρόκειται για αμαία ή όχι, αν πρόκειται για γυναίκες που ζουν στην ε, πόλη ή στην ύπεθρο Θα πρέπει λοιπόν σε, όλες, σε, τους νέες, σε όλες τις νέες να παρέχεται καθολική ε, υγειονομική περίθαλψη Και αυτό συνδέεται και με, το, με τη δεύτερη δέσμευση του Ναϊρόμπι. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η καθολική υγειονομική περίθαλψη ε, να κατευθύνεται προς ε, την ε, εξάλληψη των θανάτων βρεφών και γυναικών κατά τον τοκετό μέσω της διεύρυνσης των υπηρεσιών και της αύξησης του ε, προσωπικού που εργάζεται στον τομέα ε, της, ε, του προγεννητικού ελέγχου και του ελέγχου κατά τον τοκετό και έπειτα. Και τέλος, βία κατά των γυναικών, βία με βάση του φίλου που είναι η τρίτη δέσμευση του Ναϊρόμπιου, να δοθεί έμβαση σε μέτρα παρακολούθησης και δίωξης των επιτιθέμενων ε, ανδρών κατά των γυναικών ε, αυστηρότατα. Ε, ώστε να επιτεθούν λοιπόν όλα αυτά, καλούμε να υπάρξει χρηματοδότηση που είναι φυσικά απολύτως αναγκαία προϋπόθεση και ένας από του στόχου τη Συνόδου Κορυφής του Ναϊρόμπι θα πρέπει να είναι και η δημιουργία ενό ε, μηχανισμού που θα εξασφαλίζει τη λογοδοσία όσον αφορά την επίτευξη αυτών των δεσμεύσεων και των στόχων. Αυτά από μένα και δίνω το λόγο στον κύριο Τομπέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την κυρία Ρέγκνερ και ευχαριστώ και για την δυνατότητα να έχουμε αυτήν την κοινή συνεδρίαση. Είναι φανταστική ευκαιρία για να έχουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας. Στο σχέδιο ψηφίσματος ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στα δικαιώματα των γυναικών κοριτσιών και την ισότητα των φύλων και στις εξωτερικές της δράσεις όλος ιδιαίτερος καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ενεργά την προάσπιση των υποσχέσεών της για την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στην Σύνοδο και τις σχετικές, ε, στη σχετική της αναπτυξιακή πολιτική, την πολιτική συνεργασία. Οι διαπραγματεύσει βρίσκονται υπό εξέλιξη. Είναι λοιπόν μια μοναδική ευκαιρία να φέρουμε την ισότητα των γυναικών και την ε, χειραφέτηση των γυναικών στο κέντρο των μελλοντικών εξελίξεων είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε και επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε και τη μεθοδολογία βάσει της οποίας υπολογίζουμε πόση άμεση βοήθεια κατευθύνεται ακριβώς στον οικογενειακό σχεδιασμό. Θα πρέπει να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και στο μέλλον. Στην Επιτροπή μας, ε, στην τρέχουσα θητεία, θα δούμε πώς ε, αναλαμβάνονται οι δεσμεύσεις από την προτινόμενη Επίτροπο και πώς έρχονται και τηρώνται οι υποσχέσεις στα πλαίσια και, της, ε, και στο επίπεδο της ερχόμενης ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές που θα πάνε και στο Ναϊρόμπι και θα ξεκινήσουμε να αλλάξουμε μέλη και των δύο επιτροπών. Ξεκινάμε με ΕΛΚ ε, και ΦΑΜ και μετά πάμε στους σοσιαλιστές και ΝΤΕΒΕ και ούτω καθεξής. Η κυρία Φιτζέρελ λοιπόν πρώτη. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά να οργανώνουμε τέτοια κοινή συνεδρίαση σήμερα ε, και να είμαι εδώ. Ε, θα πρέπει να γίνεται αυτό όλο ένα και περισσότερο στο μέλλον. Διότι τα περισσότερα θέματα ξεπερνούν τα στενά όρια των αρμοδιότητων μια και μόνη επιτροπή. Ευχαριστούμε για τη δουλειά σας. Επί του ψηφίσματος που θεωρώ ότι είναι πολύ διεξοδικό, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Νομίζω ότι τα θέματα που επισημάνατε και υπογραμμίσατε και δύο είναι θέματα που με βρίσκουν σύμφωνοι. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Διεθνώς μάλιστα. Εδώ έχουμε, νομίζω, επικέντρωση διεθνή. Το καλωσορίζουμε αυτός γεγονός δεν έχω σχόλια για τις λεπτομέρειες του ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόισερ. Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία να έχουμε τις δύο επιτροπές στην ίδια αίθουσα και να μπορούμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε τι θα γίνει στο Νερόμπι. Από τη δική μα την πλευρά είναι πολύ υψηλέ οι για την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Νομίζω ότι είναι άκρο σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα του υπερπληθυσμού, για να το πω έτσι. Είναι μια σαφής δυσχέρεια και πρόκληση για τις υποσαχάριες ιδίω χώρες της Αφρικής. Για την κάθε χώρα της Αφρικανικής Υπήρου. Πραγματικά ανυπομονώ να προχωρήσουμε και να ε, αποσπάσουμε θετικά αποτελέσματα. ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και τα αποτελέσματα των συζητήσεων εκεί στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Η κυρία Ζαχαροπούλου. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την κυρία Ρέγνερ και εσένα, Τωμά, για το εξαιρετικό κείμενο που μας προτάθηκε. Ε, 25 χρόνια αργότερα δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε καθόλου τις προσπαθίες μας διότι η πρόοδος δεν είναι ποτέ κάτι το δεδομένο ως κοιόδης εισηγήτρια της ομάδας Renew θα ήθελα και εγώ να συνεισφέρω στο κείμενο και γι' αυτό θα υποβάλω μια σειρά από τροπολογίες ειδικά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία για τα κορίτσια και τις γυναίκες που είναι θύματα ε, βίας σε περιοχές κρίσης και εχθροπραξιών το συσχετισμό μεταξύ της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και την πρόσβαση στις υπηρεσίες νερού ε, και υγιεινής, ιδίω στα σχολεία, για να αντιμετωπιστεί η εγκατάλειψη από κορίτσια και η ευαισθητοποίηση ανδρών και ε, νερών αγοριών για τα θέματα αυτά, η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των ταμπού, και επίσης η ανάγκη να αναλάβει δράση η κοινωνία των πολιτών και η νεολαία της Ευρώπης στην προετοιμασία μια, ε, μιας ε, παγκόσμιας συνόδου για τον περιπληθισμό και την ε, ισότητα. Τα θέματα, τα προβλήματα παραμένουν πολυάριθμα εδώ στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φοφάνα. Ναι, εγώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ τη γραμματεία της ΔΕΒΕ και της ΦΑΜ για τη δουλειά σας, ε, για το ψήφισμα αυτό. Ε, συμφωνώ με τα περισσότερα σημεία που αναφέρεται εδώ στο ψήφισμα, δηλαδή την αναγνώριση από τις γυναίκες ότι πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο ε, και συγκατάθεση σε κάθε περίπτωση, όπως τον ελεγχόμενη άμβλωση, καθώς και τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ που ε, αφορούν το σκέλος της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Λέτε, και το αναφέρουμε, για τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, αλλά το πώς πρέπει να εργαστούμε για την εξάλληψη της κλειτοριδεκτομής και ε, το πώς πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών στην Αφρική. Ε, ημερομηνία για την στόχο, ως καταληκτήρια ημερομηνία έχουν προβλέψει το 2030. Ε, θα πρέπει επίσης να δούμε την καταστολή των γυναικών, όχι μόνο στι αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά σε όλο τον κόσμο, μαζί και την Ευρώπη. Και περιμένουμε πραγματικά με αδημονία τη, τα πορίσματα της Συνόδου του Ναϊρόμπι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κατά όλα αυτά τα προβλήματα μεταξύ άλλων την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και το πρόβλημα των πρόωρων ε, καταναγκαστικών γάμων που σε αυτή την περιοχή είναι ένα πρόβλημα μεγάλων διαστάσεων. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε το γύρο των πολιτικών ομάδων, αλλά δεν ζήτησε κανείς τον λόγο από τις ομάδες IDCR και GUE. Προχωρούμε λοιπόν με τους λοιπούς βουλευτές. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γκονσάλες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για αυτήν την πρωτοβουλία για να εργαστούμε από κοινού για θέματα τα οποία είναι πολύ ε, ε, σημαντικά έτσι ώστε να γίνουμε και χρήσιμοι για χώρες που μας χρειάζονται. Νομίζω ότι είναι μια καλή γραμμή εργασίας αυτή και θα πρέπει να προωθήσουμε και θέματα όπως είναι ε, η ε, αναπαραγωγή σεξουαλική υγεία για, γιατί στις ε, χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχει πραγματικά ε, ε, μεγάλη κινητοποίηση ε, όσον αφορά την δυνατότητα των γυναικών της Αργεντινής να αποφασίζουν για το σώμα τους και νομίζω ότι επειδή είναι μια μεγάλη χώρα η Αργεντινή μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Ε, να σας συγχαρώ λοιπόν για την ε, μέχρι τώρα εργασία και πραγματικά θα πρέπει εμείς να μεταφέρουμε, θα πρέπει μάλλον οι συνάδελφοι που θα πάνε στην ε, διάσκεψη του Ναϊρόμπι να μεταφέρουν την φωνή μας. Και πιστεύω ότι και το παράδειγμα ε, της συνεργατικής κίνησης, ε, φεμινιστικής κίνησης των γυναικών στην Αργεντινή ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό και η επίσκεψη των εκλεγμένων γυναικών της Αργεντινής τον Φεβρουάριο πραγματικά μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες και μπορεί να οδηγήσει, όπως είπα και προηγουμένως, σε αλλαγή παραδείγματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουμε η φωνή αυτών των εκατομμυρίων γυναικών που χάνουν τη ζωή τους στα πλαίσια παρανόμων αμβλώσεων. Ευχαριστούμε. Άλλοι βουλευτές θέλουν το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Γκέρενς Ρινιού. Ευχαριστώ. Άκουσα μια συνάδελφο να αναφέρει τους εξαναγκαστικούς γάμους να θυμίσω προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το κοινοβούλιο μας υπήρξε, ε, ε, ε, μου οργάνωσε αραγές με το πω. Εγώ στην προηγούμενη θητεία ήμουν ε, εισηγητής όπου με ψήφισμα ζητήσαμε να απαγορευτεί παντού κάθε εξαναγκαστικό γάμο πριν την ηλικία των 18 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι αναπτυσσόμενε χώρε, στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Προσπαθήσαμε λοιπόν στα πλαίσια των συμφωνιών μα να προβλέψουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρξει αιρεσιμότητα και με αυτή την προπόθεση προ τι τρίτε χώρε. Δηλαδή να του πούμε έχετε πρόβλημα ή θα το απαγορεύσετε βάσει νομοθεσία, οπότε παίρνετε βοήθεια ή δεν έχει περάσει νόμος ακόμα, αλλά σκοπεύεται. να περάσετε έναν νόμο, να επιτρέψετε μάλιστα να υπάρξει παρέμβαση της UNICEF και του Ταμείου του ΕΕ για τους διάφορους πληθυσμούς, επειδή δεν έχετε μόνοι σας τα μέσα να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, αλλά πρέπει να δοθεί η ευκαιρία. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη μάστιγα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι είναι έτοιμη να το κάνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει πολύ καλά το σχέδιο ψηφισματό μας και είμαι βέβαιος ότι στην επόμενη σύνοδο στο Ναϊρόμπι θα μπορέσουμε να το προωθήσουμε περαιτέρω. Την τοποθέτηση των εκπροσώπων των Ευρωπαίων πολιτών την έχουμε πάντως ε, εγκρίνει, υπάρχει και μπορείτε να την αξιοποιήσετε στις δημοτεύσεις εκεί. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλος κανείς να ζητάει το λόγο σε αυτή τη φάση. Οπότε να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε ερωτήσεις και σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήδη σε προηγούμενες συζητήσεις ε, θίξαμε τα δύσκολα στοιχεία αυτής της ε, διάσκε... αυτού του ψηφίσματος. Ε, είναι πολύ θετική, θετικό το ψήφισμα γιατί το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε όλα τα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τροχοπέδες, ξέρουμε από πού προέρχονται θα πρέπει να δείξουμε μια ισχυρή θεσμική θέση πάνω στα θέματα αυτά. Και το γεγονός ότι εσείς στέλνετε στο Ναϊρόμπι μια τέτοια ισχυρή αντιπροσωπεία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα. Και εμείς ε, στην Κομισιόν ε, έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις για το τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Επομένως, σας συγχαίρω για το ψήφισμά σας. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς με αυτό. Είναι ισορροπημένο, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα και επίσης ε, αντικατοπτρίζει και την ε, θέση της Κομισιόν όσον αφορά ε, το, το θέμα αυτό. Θέλουμε να επιμείνουμε και να υπογραμμίσουμε ε, την ε, ε, ανάγκη υποστήριξης του συστήματος υγείας. Αναφέρθηκε ε, επανειλημμένα και από εσά ε, ότι ε, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η έλλειψη πληροφόρησης όσον αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, που βασίζεται και σε στοιχεία τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα στις παραδόσεις των ε, χωρών. Πρέπει να αναπτύξουμε εργαλεία τα οποία θα μας ε, οδηγήσουν ε, σε βελτίωση της κατάστασης. Πρέπει να βασιστούμε στην ενδυνάμωση των γυναικών σε μία έρευνα η οποία δείχνει ότι στην Τινησία, το Μαρόκο, την Ποτσουάνα, την Κάνα, την Κένια, την Αιθιοπία και την Σενεγάλη, στις 7 αυτές χώρες ε, η παρέμβασή μας ε, συνδυασμένη με την βούληση των κυβερνήσεων οδήγησε ε, σε πραγματική μείωση των ποσοστών γονιμότητας. Θα πρέπει όμως να βρούμε τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά μπορεί να γίνουν αποδεκτά από τις χώρες. Επομένως, συγκεκριμένες ε, παρεμβάσεις ε, μαζί με άλλα στοιχεία, όπως ας πούμε η εκπαίδευση, είναι απαραίτητες. Επίσης, εκπαίδευση ε, σε εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων μέσα στα σχολεία ήδη. Έχει αποδειχθεί ότι η σωστή πληροφόρηση ε, μπορεί να, ακόμα και σε πιο ε, συντηρητικά περιβάλλοντα, να δώσει καλά αποτελέσματα. Εάν η πληροφόρηση ε, ξεκινήσει σωστά, αν βρει κανείς δηλαδή ένα καλό σημείο εισδοχής. το ICPD μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα, μια πλατφόρμα ε, ικανοποιητική. Ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει πισωγυρίσματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την θέση μας τόσο, ώστε να μην ε, υπάρξει ε, νέα ε, ανάκαμψη όσον αφορά και τα ε, κρούσματα σε νέους κάτω των 25 ε, ετών. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επίσης και τα αναπτυξιακά μας εργαλεία. 2,6 εκατομμύρια από το 14 ε, μέχρι το, ε, από το 14 μέχρι το 16 ε, εξ αυτών 500 και κάτι 572 εκατομμύρια The EU contribution to the Spotlight Initiative is amounting already. είναι απαραίτητα να δοθούν για την αναπαραγωγική γενική σεξουαλική υγεία. Ε, επίσης, ε, για τη ε, βία κατά των γυναικών 500 εκατομμύρια και ένα δις και ένα εκατομμύριο μόνο για το AIDS, καθώς επίσης... Of euros. And in total... Και έχουμε στο σύνολο 117 προγράμματα που αφορούν την εκρίζωση της βίας ε, ε, κατά των γυναικών και της σεξουαλικής ε, βίας. Αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το πολιτικό πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν και από πλευρά τη Κομισιόν εμεί θα είμαστε στην, στο και θα προσπαθήσουμε να διασυνδέσουμε τα όσα συμβαίνουν επί τόπου και την πολιτική πίεση που μπορεί να ασκηθεί. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για το ψήφισμα και για την υποστήριξή σας, Πρόεδρος. Εμείς σας ευχαριστούμε για τα πολύ σαφή μηνύματα. Σε αυτή τη φάση να δώσω το λόγο πάλι στην ε, Πρόεδρο Ρέγνερ για να κάνει τις καταληκτήριες παρατηρήσεις της. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας και αυτό που πρέπει να, για όλα αυτά που θα πρέπει να προσθέσουμε τεθούν και ευχαριστούμε και για την εντυπωσιακή παρέμβαση της Κομισιόν. Νομίζω ότι στην, ε, στο θα έχουμε μια εξαιρετική αποστολή που θα μπορέσει να ε, προωθήσει αυτά που πρεσβεύουμε εμείς, αυτά που έχουμε εντάξει και στο ψήφισμά μας. Λοιπόν, 26 Νοεμβρίου προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και μετά ε, ψηφοφορία των δύο επιτροπών θα γίνει στις 22-23 Ιανουαρίου του 2020 θα προσδιορίσουμε στο, στο, στο άμεσο μέλλον πιο συγκεκριμένα πια από τις δύο ημερομηνίες. Ο κ. Στομπέ, ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι η Διεθνής ημέρα κατά της βίας των γυναικών είναι 25 η Νοεμβρίου και επειδή θα έχει συνεδρίαση των επιτροπών μας ε, έως τότε, δεν θα υπάρξουν μάλλον, το σημειώνουμε τώρα, είναι, τώρα, είναι πολύ σημαντικό ε, να αναδειχθεί αυτή η διεθνής ε, ημέρα ε, διότι δυστυχώς παρατηρούμε αύξηση των φαινομένων γυναικοκτονιών στον κόσμο. Και ξέρετε ότι πρόκειται πάντοτε, πρόκειται, τα, τα, τα περιστατικά που βγαίνουν στην επιφάνεια είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, είναι χιλιάδες οι γυναίκες που δυστυχώς πεθαίνουν στα χέρια ανδρών. Ωραία, Αυτά από εμένα, λέει ο κύριος Τομπέ και συνεχίζει η κυρία ε, Ρέγνερ. Λέει ότι με αυτό μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Αποστολή των δύο επιτροπών στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για, ε, στο Ναϊρόμπι. Έχουμε τώρα μαζί μας τον συνάδελφο από ε, την συνάδελφο από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για, την, ε, για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη που είναι επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελών του συγκεκριμένου Ταμείου και θα της δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο για να μας παρουσιάσει το έργο του φορέα της. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που έχω τη δυνατότητα εδώ να συμμετέχω στην ανταλλαγή απόψεων που γίνεται σήμερα για αυτήν την σύνοδο κορυφής, εν ώψη, ε, μάλλον τη σύνοδο κορυφή στον αερόπου και να σας ε, ενημερώσω σχετικά με την έκθεση ε, για τον παγκόσμιο πληθυσμό και την ανάπτυξη που έχει τίτλο «Η επιδίωξη για ανάπτυξη και υγεία για όλους». Δεν ξέρω αν έχετε λάβει την έκθεση αυτή, έχω κάποια αντίγραφα εδώ. Εδώ σε αυτή την έκθεση αναδεικνύονται τα εμπόδια ε, και οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Το 2019 αποτέλεσε ορόσημο όσον αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Είναι η πεντηκοστή η από τη δημιουργία του Ταμείου για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και ε, η 25η επέτειος επέτειος της Συνόδου του Καΐρου για το θέμα αυτό. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, οι ομιλητές την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η σύνοδος στο Ναϊρόμπι. Έχουμε αγωνία, ξέρετε. Είναι μια σύνοδος κορυφής την οποία συγκάλεσαν οι κυβερνήσεις της Κένιας και της Δανίας και το Ταμείο ε, και στόχος είναι να δοθεί συνέχεια όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Ταμείο. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο από το 1994, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν. Να σα πω κάποια λόγια για, το, για την ιστορία του ICPD και τι ελπίδε μα ε, για τον Ναϊρόμπι. Βλέπετε εδώ στην οθόνη το 1969. Ήταν μια περίοδος κοινωνικών αναταραχών παντού, αλλά ιδίως στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ. Και πολλά από τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε σήμερα, ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών, σε έναν βαθμό τουλάχιστον πηγάζουν από τους αγώνες που έγιναν εκείνη την περίοδο. Πολύ μεγάλη πρόοδος λοιπόν έχει γίνει έκτοτε όσον αφορά την σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα. Το 1969 επίσης ήταν και μια περίοδος πανικού σχετικά με την ταχεία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Και πράγματι, το 1969 ο παγκόσμιος πληθυσμός ε, αυξανόταν ε, πιο, με, με, με μεγαλύτερους ρυθμούς από, το, από ποτεδήποτε άλλοτε στην ανθρώπινη ιστορία. Εκείνη την περίοδο η κάθε γυναίκα έφερε στον κόσμο περίπου πέντε παιδιά. Στις αναπτυσσόμενες δε χώρες έξι. Οι αριθμοί αυτοί έχουν ε, ε, μειωθεί στο μισό. Στα 17 χρόνια λοιπόν αυξήθηκε ο παγκόσμιος πληθυσμός κατά ένα δισεκατομμύριο άτομα. Ο φόβος λοιπόν ότι η αύξηση του πολιτισμού θα μπορούσε να μετριάσει τα επιτεύγματα και τα ωφέλη από την οικονομική ανάπτυξη ξεκίνησε, ε, ξεκίνησαν διάφοροι να αναλαμβάνουν δράση μέσω, για παράδειγμα, ταμείων υποτροφιών για να μελετηθούν καταρχάς αυτά τα φαινόματα. Ε, σε κάποιες, δράσ, σε κάποιες χώρες ανα, η πρωτοβουλία να δημιουργηθούν υπηρεσίες οικογενειακού σχεδιασμού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε, σε γυναίκες, ε, εφόσον το επιθυμούσαν, να παρατείνουν ε, ή να αναβάλουν τη δημιουργία οικογένειας. Επίσης ενθαρρύθηκαν ζευγάρια να ε, μειώσουν τα παιδιά που έχουν ή να, μην κάνουν και καθόλου παιδιά. Το, το, τη δεκαετία του 80 αυξήθηκε η διαθεσιμότητα αντισυλληπτικών και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ αναπτύχθηκαν και νέες τεχνολογίες αντισύλληψης ε, οι οποίες διεύρυναν τις επιλογές για ζευγάρια και για γυναίκες. Όμως, Παρά το γεγονό ότι η ποικιλία και η ποσότητα των αντισυλληπτικών αυξήθηκαν, πολλές ε, γυναίκες εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια. Εμπόδια κοινωνικά, θεσμικά, οικονομικά, πολιτισμικά, τα οποία τις εμπόδιζαν από, τον, από την πρόσβαση σε πληροφόρηση και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να τι βοηθήσουν να, ε, να αποφασίσουν εκείνε για τον οικογενειακό σχεδιασμό τους. Επίσης, γυναίκε σε όλο τον κόσμο ε, άρχισαν να ισχυρίζονται ότι δεν ήταν μόνο η γονιμότητα αυτή που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, αλλά μια σειρά από ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ε, τα οποία θα πρέπει, στα οποία θα πρέπει να δοθεί η αναγκαία προσοχή. Στη δεκαετία του 80 και του 90 πολλές οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, ιδίω οργανώσεις γυναικών, ζητούσαν την αντικατάσταση των προγραμμάτων οικογενειακού σχεδιασμού που στην ουσία ε, κατά βάση ε, έδιναν αντισυλληπτικά γυναίκες ε, με μια ευρύτερη προσέγγιση και αντίληψη ότι θα πρέπει το βασικό, ο βασικός γνώμονας να είναι τα δικαιώματα των ε, γυναικών και όχι απλά ε, δημογραφικά κριτήρια. Και έτσι ο οικονομικός σχεδιασμός αποτέλεσε μόνο ένα μέρος της συνολικότερης πολιτικής ε, που θα, πρέπει, που θα έπρεπε να χαραχτεί για την εξασφάλιση σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας όλου του πληθυσμού. Αυτά όλα συνέβαλαν στην ε, προετοιμασία της ε, Συνόδου Κορυφής του 1994 και πραγματικά οδήγησαν σε μια μεταστροφή όσον αφορά την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων που αναγνωρίζουν πλέον ότι οι ατομικές και οι συλλογικές ε, επιδιώξεις μπορούν να συμφιλειωθούν υπό, το, τη σκέπη ολοκληρωμένων πολιτικών. Βεβαίως ε, για να επιτευχθεί ανάπτυξη χρειάζεται να παρακολουθείτε και η, η δημογραφική διάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει ταυτόχρονα να προωθούνται και η, να προωθείται η λήψη αποφάσεων εξατομικευμένων από μεμονωμένες από την κάθε γυναίκα ξεχωριστά. Και θα πρέπει η, τα δικαιώματα της, της γυναίκας να είναι ο γνώμονας για την ανάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών. Και αυτό που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις ήταν να δοθούν στις, γυ... στις γυναίκες και στα ζευγάρια μια σειρά από υπηρεσίες οικονομικού σχεδιασμού που και να αναλυφθούν οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερη ισότητα των φύλων. Αυτό ήταν και πραγματικά το πρώτο, ε, ο πρώτος στόχος. 2015. Ατζέντα 2015 30 και βιώσιμη, στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου ρητός αναγνωρίζεται η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ως ανάπτυξη που θα συμβάλλει στην ισότητα των γυναικών. Έχουμε συγκεκριμένα το στόχο 3 ε, για την ε, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τον στόχο 5 για την ισότητα των φύλων. Οι υπηρεσίε οικογενειακού σχεδιασμού επίσης ε, εντάσσονται ε, στην παρακολούθηση που γίνεται όσον αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων και αντίστοιχη δουλειά γίνεται και από την Κομισιόν για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Οι SDG αναγνωρίζουν την ανάγκη να υπάρχει καθολική υγειονομική περίθαλψη που θα πρέπει ε, να καλύπτει ε, τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα της ζωής τους. Όπως ε, και η ICPD, έτσι και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ε, ε, υποστηρίζουν και υπογραμμίζουν την ισότητα όσον αφορά όλους τους στόχους αυτούς. Γιατί μιλάμε ακόμα για αυτή τη διάσκεψη 25 χρόνια μετά. Ποια διαφορά έκανε. Νομίζω ότι έκανε μεγάλη διαφορά πάνω από 40% ε, έπεσε το ποσοστό θνησιμότητας ε, και κατά ένα ε, τρίτο των γυναικών που είχαν παντρευτεί πριν από την ηλικία των 18 ετών έπεσε σημαντικά Επίσης, 10% ε, αύξηση στις ε, ε, γυναίκες που είναι παντρεμένες, αλλά και που χρησιμοποιούν προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ σωστά. Δηλαδή, ε, ε, ο ρυθμός είναι πάρα πολύ αργός ε, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε δει ότι δεν υπάρχει αρκετή η ταχύτητα έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το, 1900, το 2030. Επίσης εξακολουθούν ε, να είναι εκατομμύρια αυτοί οι οποίοι δεν ε, ε, απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων του όσον αφορά τη εκλογική και αναπαραγωγική υγεία. Κυρίως πρόκειται για γυναίκες που ζουν σε μη περιοχέ περιοχές και οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

στις ε, χώρες για τις οποίες έχουμε, ε, τα, ε, έχουμε στοιχεία, μονάχα το μισό, των, το 50% των γυναικών λένε ότι έχουν κάποια πρόσβαση σε προγράμματα σεξουαλικής υγείας. Δεν έχουν μειωθεί επίσης οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των νεογνών που έχουν πρόσβαση πρόσβαση σε ε, ε, ε, περίθαλψη υγείας αμέσως μετά την γέννησή τους. Το γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι εδώ που είμαστε τώρα, προφανώς δεν ήταν εύκολο. Μερικές φορές τα εμπόδια ήταν οικονομικά, άλλες φορές αφορούσαν τις κοινωνικές δομές που επιτρέπουν στους άντρες να έχουν όλη την εξουσία. Ε, πέρα από αυτά πάντως ε, υπάρχει μεγάλη συνένεση ότι όλοι οπουδήποτε θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ε, πληροφορίες και οπωσδήποτε περίθαλψη όσον αφορά την αναπαραγωγική και σεξουαλική τους υγεία. Τα τελευταία χρόνια ε, είδαμε επίσης ε, και μία αναζωπήρωση της προσοχής όσον αφορά ε, την δημογραφική αλλαγή. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει και το, η δυνατότητα να ε, να έχουν αυτό το δημογραφικό μπόνους ε, λόγω των πολλών νέων με ταυτόχρονη μικρή, μικρό ποσοστό εγκυμοσυνών. Βεβαίως, ε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες μπορεί να είναι αναπτυγμένες αλλά έχουν πολύ μικρό ποσοστό γονιμότητας πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά κοινωνικά κλπ ε, ε, ε, λόγω του γυράσκοντος πληθυσμού. Ε, οποιασδήποτε προσπάθειες ε, τροποποίησης ε, βέβαια των δημογραφικών τάσεων με απότομο τρόπο και επεμβατικό θα πρέπει να αποφεύγονται καθότι ελοχεύει ο κίνδυνος παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων. Οι κοινότητες και οι κυβερνήσεις οφείλουν οφείλουν να συλλέξουν στοιχεία ε, τα οποία θα ε, καλύπτουν ε, την αντιμετώπιση αλλά στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ολοκληρώσω εδώ. Sorry. I, I, didn't want to take so long, but it really, there is some history Ναι, κοιτάξτε, μερικά ιστορικά στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνει κανείς προς τα που πάμε αν δεν ξέρουμε το παρελθόν. Άρα πολλά ε, πράγματα μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Οχτώ γυναίκες πεθαίνουν κάθε μέρα ε, από λόγους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Ε, και πολλές είναι οι γυναίκες οι οποίες κάποια στιγμή της ζωής τους θα αντιμετωπίσουν κάποια πράξη βίας. ο στόχος ή μάλλον η στόχη της διάσκεψης του Ναϊρόμπι είναι ε, να επιταχύνουν και να ε, εφαρμόσουν πλήρως τα όσα είχαν αποφασιστεί το 1994. Ε, είναι, υπάρχει ένας ευρύς ε, συνασπισμός ανθρώπων που πραγματικά επιθυμούν να υλοποιηθεί αυτό το ε, θεματολόγιο. η διάσκεψη του Ναϊρόμπι εστιάζει σε πέντε θέματα τα οποία σας δείχνω εδώ. Ε, ε, είναι στοιχεία τα οποία αποσκοπούν στην περίθαλψη, την κάλυψη της υγείας, ε, στα προγράμματα δράσης για την επικύρωση των όσων επιτευγμάτων έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα, ισότητα ανδρών γυναικών, απάλληψη της βίας κατά των γυναικών κλπ όλοι εδώ, αλλά ε, κυρίως ε, και οι βουλευτές ε, που θα είναι στην αντιπροσωπεία του Ναϊρόμπι, παρακαλώ, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Ε, και ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο και αν πραγματικά είμαστε ε, εξαιρετικά ευχαριστημένοι για την σύγκληση της διάσκεψης του Ναϊρόμπι, πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια όλων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο σας. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται παρεμβάσεις από τα μέλη, αλλά από την, οργάνωση για τον, την Παγκόσμια Οργάνωση για τον Οικογενειακό Σχεδιασμό. κυρία Ράιτ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που μου δίνετε και το λόγο και συγχαρητήρια για την κοινή σας συνεδρίαση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το είδος τη συνεργασία. Εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο του τη Ομοσπονδία μα για τον οικογενειακό σχεδιασμό. Εργαζόμαστε σε πολλά κράτη για τα θέματα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Ω Ευρωπαϊκό Δίκτυο έχουμε πολλά κράτη-μέλη στην Ευρώπη και Κεντρική Ασία για να βεβαιωθούμε ότι οι νέοι μπορούν να ζουν με προστασία των, των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και αλλού δεν έχουμε ε, όρια και δεν γνωρίζουμε σύνορα στη δράση μας ε, και υπάρχει και ένα σχετικό διεξοδικό πρόγραμμα δράσης. Πιστεύουμε ότι η σύνοδος του Ρουμπή για την 25η επέτειο του προγράμματος δράσης είναι μια κρίσιμη ευκαιρία. Πρέπει να δείξουμε την πολιτική μας βούληση και τις οικονομικές ε, δεσμεύσεις μας να τις κάνουμε πραγματικότητα. Η σύνοδος είναι μια ευκαιρία να συμπληρώσουμε και να υποστηρίξουμε τι πραγματικέ πρωτοβουλίε του ΙΕ που έχουν λάβει χώρα σε όλε τι περιοχέ του κόσμου Φέτο. Αξιοποιώντα την ευκαιρία να πιέσουμε τι κυβερνήσει να αναλάβουν δεσμεύσει. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να καλέσει ας πούμε, με τη σειρά του την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματο δράση και να τηρήσουν ή να διατηρήσουν την μακροχρόνια υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε λοιπόν το κοινό ψηφίσμα των Επιτροπών ΔΕΔΕ και ΦΑΜ και ελπίζουμε θα το υποστηρίξουν και οι ευρωβουλευτές. Ε, μερικά σχόλια. Υποστηρίζουμε την έκκληση του Ευρωκοινοβουλίου για σαφή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σεξουαλικά και ευρωπαϊκά δικαιώματα των γυναικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο τα τελευταία χρόνια που μόλις σας παρουσίασα, ακούσαμε ότι πολλά παραμένουν ημιτελή. Η οικονομική φραγμή είναι ε, διαρκώς αντινόμενη σε ένα πλαίσιο που δεν επιτρέπει την ε, πολιτική πρόοδο. Γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μέλη της να παίξουν έναν ενεργότερο ρόλο ώστε να προωθήσουν τα δικαιώματα που κι εμείς προσπιζόμαστε από οικονομική και δημοσιονομική άποψη. Πραγματικά πρέπει να υπάρξει ένα πολύ ε, αυστηρό σύστημα λογοδοσίας, ελέγχου της ανάληψης υποχρεώσεων, που να ξεκινήσει από τον Αρόμπι. Νομίζω πραγματική δουλειά θα ξεκινήσει μετά τη Σύνοδο και θα δείξουμε κατά πόσο είμαστε πιστοί στις υποσχέσει μα και στα λόγια μα. Η επικέντρωση Στου τρει στόχου που αναφέρατε είναι σημαντικό. Εμεί εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών, κοιτάζουμε την υλοποίηση του προγράμματο δράση και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιδιώξουμε του κατάλληλου στόχου. Ελπίζουμε ότι ο χώρος που θα προσφερθεί στην κοινωνία των πολιτών θα επιτρέψει την πραγματική ε, υλοποίηση του συστήματος για μια συνολική ε, αλλαγή στην νοοτροπία και την εκπαίδευση των σε σχέση με τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγική υγείας. Μιλάμε για παρεμελημένες ε, προτεραιότητες, ενώ έχουμε τη μεγαλύτερη γενιά αριθμητικά σε νέους. Πρέπει να ε, ενέσουμε επίσης την επικέντρωση του ψηφίσματος σε αξίες και την ανάγκη αλλαγή της νοοτροπία ε, σε επίπεδο οικογενειών αλλά και στο πολιτικό κλίμα τη σημερινή εποχή. Κάθε άτομο στην Ευρώπη και εκτό θα πρέπει να έχει ασφαλή και υγιή αναπαραγωγική σεξουαλική ζωή. Πιστεύουμε επίση ότι είναι κρίσιμη σημασία να γίνουν ε, οι σωστοί συσχετισμοί. Το είπα ήδη αλλά το πρόγραμμα δράσης αυτό και άλλα διεθνή πλαίσια, όπως η Ατζέντα για το 2030 ή η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, που θα γιορτάσει την 20η της ε, επέτειο το 2020. Όλα αυτά είναι σημαντικά για να πετύχουμε τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης 3 για την υγεία και 5 για την ισότητα των φύλων στην ε, χάρτα θα πρέπει να εμπνευστούμε από την ολιστική προσέγγιση που συστήνεται για τα δικαιώματα των γυναικών όπως προβλέπει και το πρόγραμμα δράσης πλατφόρμα για το Πεκίνο ε. αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Πεκίνο ΣΥΝ 25 και τους σχετικούς ε, στόχους του πρόγραμματος βιώσιμης ανάπτυξης. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν σε όλε τι χώρε τα θέματα αυτά, καθώ και στα επίπεδο τη αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι σημαντικό το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου να καλύψει ε, το τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτε χώρε, αλλά και στην κατάσταση εντό Ευρώπη. Υπ' αυτήν την έννοια, το ψήφισμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει εκκλήσει για μια ισχυρότερη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την κύρωση και την έγκριση τη ε, Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, πιστεύουμε ότι είναι εξίσου σημαντικό το ψήφισμα να αναγνωρίσει την πραγματική παγκόσμια προσταδρόμηση στην προστασία των δικαιωμάτων των γενικών. Και εδώ θα πρέπει να προστατεύσουμε σε αυτό το πλαίσιο και του προσπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι σχετικέ οργανώσει. Και πολιτικώ, αφήνοντα να υψώσουν τη φωνή του, και οικονομικώ καταστολή ε, περιορίζει την ε, ελευθερία των γυναικών παντού αλλά και στην Ευρώπη. Περικοπές στην προστασία των ε, σεξουαλικών και απαραγωγικών δικαιωμάτων παρατηρούνται και εκτός Ευρώπης και εντός. Θα πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουμε τις αρχές της ισότητας των φίλων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε και ελπίζουμε θα συνεχίσουμε την επικοδομητική μας συνεργασία καταλήγοντας σε ένα πολύ ισχυρό ψήφισμα. Ευχαριστώ σα ευχαριστώ όλους. Οι πληροφορίες που μας δώσατε είναι πολύ χρήσιμες για τους συναδέλφους που θα πάνε στη Σύνοδο την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά πριν δώσω το λόγο στην συμπρόεδρο Ρέγνερ, να πω ότι έχουμε μια ομάδα επισκεπτών εδώ που κάλεσαν, κάλεσε ο κύριος Νόιζερ από μη κυβερνητική οργανώσεις από το Voice of Audit Foundation